El señor presidente. Queridas amigas y queridos amigos, buenas noches. Reanudamos la. Καλησπέρα σας. Ξεκινώ μια ανακοίνωση. Οι Βρετανικές Αρχές με ενημέρωσαν για την ε, αντικατάσταση της κυρίας Wallace από την κυρία Ερβέκα Elizabeth Taylor από την 8η Μαρτίου 2012. Καλωσορίζω την νέα συνάδελφο με βάση τον κανόνα του άρθρου 3 παράγραφος 2 εκρεμεί η επαλήθευση της διαπίστευσης της Έσω του κυρία Τέιλορ μπορέσει να παρακαθίσει στις συνεδριάσεις μας. Μένει να επιβεβαιωθεί ότι δεν ε, κατέχει